Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι, φοβάμαι ότι θα αρχίσουμε από το σημείο 5. θα επανέλθουμε στις συνήθειες εργασίες της Επιτροπής ΕΛΕΦ ΛΥΜΠΕ Τελείωσε η συνεδρία των συντονιστών και ξαναρχίζει τώρα η κανονική μας δουλειά. Το θέμα που αφορά το πρόγραμμα των δικαιωμάτων των πολιτών. Η πρώτη, ο πρώτος τριμερής διάλογος είχε αρχίσει 4 Δεκεμβρίου, έγινε και ο δεύτερος, ο τρίτος προγραμμα, προβλέπεται για τέλη Φεβρουαρίου και τώρα θα ακούσουμε την συγκήτρια κυρία Γκόντς Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπατε, έγιναν ήδη δύο τριμερείς διάλογοι και περιμένουμε ακόμη έναν στις 18 Φεβρουαρίου και έναν τέταρτο 15 Μαρτίου. Συμφωνήσαμε να αλλάξει ο τίτλος από την αρχή, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για μας. Υπήρχαν μερικές διαφωνίες σε συγκεκριμένα άρθρα και σημεία συζητήθηκε το αν θα χρησιμοποιηθεί η γλώσσα και η ορολογία της συνθήκης ή της χάρτας και τώρα ψάχνουμε έναν συμβιβασμό δηλαδή η γλώσσα της χάρτας στην εξηγηματική έκθεση, στην αιτιολογική έκθεση σαν να λέγαμε μέσα σε αγγίλες γιατί γενικότερα το κοινοβούλιο χρησιμοποιεί περισσότερο την ορολογία της χάρτας. Το επεξεργαζόμαστε λοιπόν για τα προγράμματα καινοτομίας και κοινωνικής περίθαλψης υπάρχουν μερικά προβλήματα. Ε, ε right και για τα θέματα δικαιωμάτων των καταναλωτών επίσης ε, ακόμα δεν έχει λυθεί το θέμα. Εμείς θα θέλαμε να διατηρηθούν αυτές οι ρήτρε. Συζητήσαμε πολλά άρθρα και σημεία, δεν αποφασίσαμε ακόμα τον τελικό συμβιβασμό. Υπάρχει και ένα θέμα που πρέπει μαζί να λύσουμε, το θέμα τον κατά, κατά κατεξουσιοδότηση πράξεων στο πρόγραμμα Justice. Και πρέπει εδώ να φτάσουμε σε κάποια εναρμονισμένη θέση για να μην έχουμε κάθε φορά διαφορετική διατύπωση και θέση με κάθε θέμα που τίθεται. Μήπως θέλει κανείς να σχολιάσει αφού ακούσαμε τη σύνοψη της εισηγητρίας κυρίας Γκάντς, αν όχι, περνάμε στο επόμενο σημείο, το 10, όπου η εισηγητής είναι η συνάδελφός μας κυρία Άννα Χέντ. Θα ακούσουμε και την παρουσίασή της και τα σχόλια της Κομισιόν της κυρίας Μπερέντα από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων. Ορίστε. Κύριο Μπερέντα. Ευχαριστώ. Η πρόταση που εξετάζεται αφορά τροποποίηση του υπάρχοντος κανονισμού για τις πρόδρομες ουσίες ναρκωτικών Πολλές φορές υπάρχει θεμητή χρήση τους, αλλά μπορεί να υπάρξει και κατάχρηση για την παραγωγή παρανόμων ναρκωτικών. Και αυτή τη στιγμή αυτό που ισχύει είναι ότι παρακολουθούμε το εμπόριο, την εμπορία τους αρκετά αυστηρά. Το 2009 κάναμε μια αξιολόγηση της λειτουργίας του ισχύοντος κανονισμού με βάση το γεγονός ότι υπήρχε πολύ, είχαν πολύ ψηλ, πάρα πολλές προσπάθειες ε, κατάχρησης ε, μια συγκεκριμένη ουσία του οξικού ανιδρύτη. Πράγμα που μας οδήγησε και σε επικρίση α, οδήγησε σε επικρίση από το Διεθνές Συμβούλιο Ναρκωτικών που βασίζεται στη, στα κείμενα του ΟΗΕ διαπιστώσαμε ότι γενικά ο κανονισμός και το καθεστώς εποπτείας λειτουργούν σωστά, αλλά υπάρχουν και ορισμένες αδυναμίες ιδιαίτερα για αυτή την ουσία του οξικού ανιτρίτη. Υποβάλαμε την έκθεσή μας στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, την αξιολόγησή μας δηλαδή. Το Συμβούλιο δέχτηκε συμπεράσματα που ζητούν από την Κομισιόν να προτείνει τροποποίηση του κανονισμού για να λυθούν και αυτά τα θέματα ελήψεων στον κανονισμό το Κοινοβούλιο δεν είχε ακόμη εγκρίνει. Κάναμε λοιπόν μία πολύ λεπτομερή μελέτη αξιολόγησης για να δούμε πώς θα μπορούσε να τροποποιηθεί ο κανονισμός με διαβούλευση όλων των ενδιαφερομένων εταιριών, βιομηχανικών τομέων και ιδίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι επιλογές πήγαιναν από το 0 μέχρι σε αυστηρότερα μέτρα και απαγορεύσεις. Και από εκεί προταυτίσαμε την καλύτερη επιλογή που θα ήταν η υποχρέωση του τελικού χρήστη του όμικρον α να γράφει, να καταγράφει κάθε χρήση. Και οι εταιρείες που πολλούν οξικό ανιδρύτη πρέπει να καταγράφουν τις πωλήσει, αλλά όχι οι εταιρείε που τον χρησιμοποιούν για να δημιουργήσουν άλλες ουσίες με βάση αυτόν. Εκτός από αυτή την ρήτρα, αυτό το μέτρο, προτείνουμε επίσης και τον καθορισμό, τη δημιουργία μιας τράπεζας δεδομένων που να διευκολύνει την πληροφόρηση που απαιτείται ήδη από χώρες μέλη για περιπτώσεις κατασχέσεων για χρήση που υποπτευόμαστε ότι θα είναι παράνομη και καθορισμό καταλόγου όλων των τελικών χρηστών και εμπορευομένων που πράγμα που θα διευκολύνει την επαλήθευση από τις χώρες μέλη της πραγματικής χρήσης των προδρόμων αυτών. Και τέλος, τελευταία αλλαγή που ακούσατε και στο προηγούμενο θέμα, αλλάξαμε τους κανόνες της επιτροπολογίας για τις κατεξουσιοδότησης πράξεις για να συμφωνούμε με τη συνθήκη της Λισαβόνας άλλες μικρότερες αλλαγές που ίσως δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε σήμερα, αλλά υπάρχουν, αν θέλετε θα σας τις αναφέρω. Τέλος, υπάρχει και δεύτερη πρόταση για τους προτρόμους ναρκωτικών που τη συζητάει η Επιτροπή Ίντα και αφορά το εξωτερικό εμπόριο των ε, προτρόμων ναρκωτικών και με αυτό ασχολείται η Γενική Διεύθυνση Τελωνιακών Θεμάτων και το Συμβούλιο θα την εξετάσει επίσης. Εκείνη της πρότασης το περιεχόμενο δεν αφορά άμεσα το δικό μας θέμα εδώ, αλλά την αναφέρω γιατί υπάρχει και θα συνσυζητηθεί με το δικό μας θέμα. Ευχαριστούμε. Η εισηγήτρια κυρία Χέντ θέλει να μας παρακάνει την παρουσίασή της. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω όμως σου ειδικά και γι' αυτό ίσως χρειαστούν τα ακουστικά σας και οι διερμηνείς. Η Κομισιόν έκανε μια δήλωση που εξηγούσε το περιεχόμενο της πρότασής της δεν θα επισέλθω λοιπόν εδώ σε λεπτομέρειες. Υπάρχουν ήδη διατάξεις για τον έλεγχο και την εποπτεία της εμπορίας των προδρόμων ναρκωτικών που λειτουργεί μέχρι τώρα ικανοποιητικά και βασίζεται σε σύμβαση του ΙΕ. Σήμερα μιλούμε για τεχνικές αλλαγές προς τον ισχύοντα κανονισμό, δηλαδή για θέμα τελείως τεχνικό. Με την πρόταση αυτή πάντως θέλουμε να προσαρμοστούμε, να προσαρμοστεί η ισχύουσα νομοθεσία και με την συνθήκη της Λισαβόνας, δηλαδή για τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας ουσιών, ιδιαίτερα του οξικού ανιδρύτη, που χρησιμοποιείται για την παρασκευή παραγωγή ηρωίνης. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να μην φτάνει σε λάθος χέρια η ουσία αυτή για την παραγωγή δηλαδή παρανόμων ναρκωτικών. Η Κομισιόν αρχίζει με τις κατεξουσιοδότηση πράξεις και βασίζεται και αυτό νομίζω είναι σωστό. Αλλά βέβαια θα συζητηθεί κατά τον τριμερή διάλογο που προβλέπεται. Η Κομισιόν μίλησε και για λεπτομέρειες που θα τις συζητήσουμε σε άλλη φάση και θα τις δω και εγώ στην έκθεσή μου, κυρίως την καινούρια τράπεζα δεδομένων, πανενοσιακή τράπεζα δεδομένων που προτείνεται, για να, με στόχο να δημιουργηθεί επαρκής προστασία τα κράτη-μέλη λοιπόν θέλουν να καταπολεμηθεί η κατάχρηση αυτών των προδρόμων που θα στοχεύει βέβαια την παραγωγή παρανόμων ναρκωτικών. Επίσης μιλάει η Κομισιόν για εξαιρέσεις για πολύ μικρές εταιρείες που δεν θα απαιτείται να εγγράφονται σε μητρώα για την χρήση του ομικρονάλφα. Θα συνεννοηθώ λοιπόν με τους Κιώδης και με την Κομισιόν και με οποιονδήποτε συνάδελφο ενδιαφέρεται και με χαρά θα ακούσω τυχόν σχόλια των Σκιωδών ιδίω. Ευχαριστώ κυρία Χέντ. Ας μας μιλήσουν τώρα οι Σκιώδης ηγητές. Πίρκερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Διαπιστώνω πρώτον ότι δυστυχώς η πολιτική καταπολέμηση των ναρκωτικών ε, δεν είναι όλο και περισσότερο διαφεύγει του κέντρου της προσοχής μας. Η συζήτηση που κάνουμε τώρα, οι τροπολογίες που αφορούν την καταγραφή σε Μητρώα για τις πρόδρομες ουσίες, είναι όμως ένα στοιχείο που θα πρέπει να επαναφέρει στο κέντρο της προσοχής μας ε, τα θέματα αυτά. Διότι, όπως ξέρετε, δεν έχει μειωθεί η κατανάλωση ναρκωτικών. Αντίθετα, ε, τρέπεται προς άλλες ουσίες και μάλιστα αυξάνεται. Γι' αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε η στρατηγική μας και οι διατάξεις μας να επανεξετάζονται από καιρούς καιρό και να προσαρμόζονται στις νέες πραγματικότητες. Ο κανονισμός αυτός και η πρόταση για μια τροπολογία, αυτό το στόχο έχει, υποστηρίζω αυτή την πρόταση της Επιτροπής, κατηγορηματικά και τις προτάσεις της συγκήτριας ούτως ώστε αυτή η ουσία, ο μικρον α, να σημαίνει υποχρεώσεις και τον τελικό χρήστη, γιατί εδώ υπάρχουν τα προβλήματα. Δεν αρκεί μόνο η παραγωγή να καταχωρίζονται, εφόσον δεν ξέρουμε τι ποσοστό των ουσιών εκτρέπεται του ε, νομίμου στόχου κατά τη διάρκεια της εμπορίας. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει αυτή η υποχρέωση. Σωστά τονίσατε ότι αυτή η πρόδρομη ουσία, όπως και άλλες παρόμοιες, χρησιμοποιείται για νόμιμες χρήσεις, ε, για υπολογιστές. Τις χρειαζόμαστε αυτές τις ουσίες λοιπόν για άλλες χρήσεις. Όμως αυτές οι ίδιες ουσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την ε, παραγωγή ηρωίνης. Πρέπει λοιπόν να περιορίσουμε τη χρήση της, να πολεμήσουμε την εγκληματικότητα που σχετίζεται με την εμπορία ηρωίνης και γι' αυτό υπάρχει αυτή η υποχρέωση καταχώρησης για τους τελικούς χρήστες. Υποστηρίζω λοιπόν αυτή την κατεύθυνση. Υποστηρίζω τις τροποποιήσεις της υποχρέωσης καταχώρησης. Τη δημιουργία λοιπόν αυτής της βάσης δεδομένων για αυτές τις ουσίες Εξετάζοντας τις διάφορες εναλλακτικέ που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρώ ότι η πέμπτη εναλλακτική λύση είναι η πιο εφικτή. Όπου θα λαμβάνονται υπόψη, θα συντάσσονται καλύτερα και ε, μελέτες ε, σχέσεις κόστους αποτελέσματος. Προτιμώ λοιπόν αυτήν την ε, επιλογή 5, γιατί νομίζω ότι είναι η πιο εφαρμόσιμη λύση. Και έτσι νομίζω το αντιμετωπίζουν και οι ενδιαφερόμενοι φορεί. Και θα έχουμε δυνατότητα να κάνουμε έναν αποτελεσματικό έλεγχο. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Υποστηρίζω πλήρω τι προτάσει τη Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον εισηγητή. Δύο ερωτήσει στην Επιτροπή για αυτή την πρόταση. Πώς αποτιμάτε την αναλογικότητα της πρότασης, όπως είπε και ο κύριος Πίρκελ. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, άτομα που για, νόμιμους, ε, για νόμιμες χρήσεις χρησιμοποιούν αυτήν την ε, ουσία και το ποσοστό της χρήσης που αφορά την ηρωίνη είναι πολύ μικρό. Θα ήθελα να μάθω πόσες επιχειρήσεις θα χρειαστεί τώρα να παίρνουν άδεια, να εγγράφονται στα Μητρώα, αυτό δεν θα δημιουργήσει καθυστερήσει για τι εταιρείε, γιατί πρέπει να εγγραφούν σε κάποιο μήτρο, να εγκριθεί η εγγραφή τους κτλ. Αυτό δημιουργεί καθυστερήσει. Και επίση, τι επιπτώσεις θα έχει αυτή η πρόταση για τους χρήστες ηρωίνης. Γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα με τη χρήση της ηρωίνης είναι ότι αυτοί που την κατασκευάζουν, ε, την ε, ε, κάνουν μείγματα μετά με πολλές ιδιαίτερα τοξικές ε, ουσίες, ε, δηλητήρια. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε αν έχετε μια εκτίμηση για αυτό το θέμα. Επίσης στην πρότασή σας λέτε ότι μειώθηκε ο όγκος αυτής της ουσίας που κατασχέθηκε από το 2008 και εντεύθεν. Θα ήθελα να μας πείτε κατά πόσο μειώθηκε και γιατί μειώθηκε παρακαλώ. Επίσης, έχουμε μια γνωμοδότηση με πολλά σχόλια από τον αρμόδιο για την προστασία των δεδομένων. Ε, πώς σχολιάζετε τα δικά του σχόλια αναφέρει συγκεκριμένα ότι ορισμένα πρέπει να είναι στο κυρίω κείμενο, όχι στο παράρτημα. Επίσης αναφέρει ποια συγκεκριμένα στοιχεία πρέπει να καταχωρίζονται για να μην καταχωρίζονται προσωπικά δεδομένα ευαίσθητα. Αυτό δεν το κάνετε εσείς μέχρι τώρα. Επίσης, τι εννοείτε όταν μιλάτε για την ε, καταλληλότητα και ακαιρεότητα του ε, ετούμενου εγγραφής ε, στο Μητρό. Πώς θα τα αποτιμάτε όλα αυτά. Πολλές ερωτήσεις λοιπόν θα ήθελα να απαντηθούν. Ίσως θα ήταν χρήσιμη ε, μια απαρίθμηση των τομέων της οικονομίας όπου χρησιμοποιείται αυτή η ουσία. Θα ήταν σκόπιμη για να ε, διαμορφώσουμε άποψη για το θέμα αυτό και ευχαριστώ. Έλεγα λοιπόν, θέλει να αντιδράσει η Επιτροπή και μετά θα στραφούμε για τελικά σχόλια προς ε, την εισηγήτριά μας, η Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και την κυρία Χέντ και τον κύριο Μπέρκα για τα γενικά πολύ θετικά σχόλιά τους και την ε, στήριξη που εξέφρασαν για μια σειρά από τις προτινόμενες διατάξεις. Τώρα για τις ερωτήσεις της κυρίας Κέλλα. Βεβαίως, κάναμε μεγάλη προσπάθεια και αφιερώσαμε πολύ χρόνο στην αποτίμηση της αναλογικότητας και της ε, ε, αποτελεσματικότητας που θα έχει η δράση μας σε σχέση με το κόστος που οπωσδήποτε θα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις. Θα δείτε στην μελέτη επιπτώσεων πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, αριθμητικά στοιχεία. Φυσικά είναι πάντα εκτιμήσεις. Θεωρούμε λοιπόν ότι σε όλη την Ένωση θα χρειαστεί να εγγραφούν γύρω στις 2.500 επιχειρήσεις, αλλά μία φορά μόνο θα χρειαστεί να εγγραφούν. Δεν θα χρειάζεται ανανέωση ε, κάθε χρόνο τακτικά, εκτός αν κάποιο κράτος μέλος θεωρεί ότι θέλει να ελέγξει ή να ελέγχει ε, τα δεδομένα της εγγραφής από καιρού εις καιρών. Τώρα για τους χρήστες της ηρωίνης. Πολύ λεπτό θέμα. Πρέπει όλοι να έχουμε συνέστηση του ότι η ηρωίνη έρχεται κυρίως από το Αφγανιστάν, εκτός της Ένωσης. Αν επιτύχουμε να αποφευχθεί η χρήση στο Αφγανιστάν της ουσίας αυτής για την παρασκευή ηρωίνης, τότε οι παραγωγοί θα προσπαθήσουν να την ε, βρουν αλλού αυτή την ουσία. Στην Ινδία, την Κίνα, το Ιράν, οπουδήποτε. Εμείς ως Ένωση, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αποφύγουμε τουλάχιστον η δική μας αυτή πρόδρομη ουσία να μην πηγαίνει παράνομα στο Αφγανιστάν. Θα μειωθεί ε, η ηρωίνη στην κυκλοφορία. Το ελπίζουμε βεβαίως. Αλλά αν θα το επιτύχουμε θα εξαρτηθεί από το ότι θα κάνουν και άλλες χώρες. Εάν θα ενισχύσουν τους ελέγχους τους. Ελπίζουμε ότι αυτά τα συμπληρωματικά μέτρα της Ένωσης θα προκαλέσουν ε, συμπληρωματικά μέτρα και σε άλλες χώρες που προμηθεύουν αυτή την ουσία. Η Ένωση έχει διμερείς συμφωνίες για τις ουσίες αυτές με την Κίνα και μια σειρά από άλλες τρίτες χώρες. Βεβαίως έχει μειωθεί η κατάσχεση ηρωίνης αρκετά τα τελευταία χρόνια. Τα στοιχεία τα περιέχει η μελέτη επιπτώσεων. Το 2009 λοιπόν, για παράδειγμα, κατέβηκε σε μόνο 33 τόνους και την επόμενη χρονιά μειώθηκε ακόμη περισσότερο. Ουσιώδης μείωση. Λόγος γι' αυτό είναι ότι έχουμε συνεργαστεί πολύ στενά με τα κράτη-μέλη και με τις εταιρείες για την καλύτερη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας αυτή η μέγιστη τιμή που παρατηρήσαμε το 2008 οφείλεται και στο ότι σε κάποια κράτη-μέλη οι αρχές και οι επιχειρήσεις δεν συνεργάζονταν όσο θα έπρεπε και δεν είχαν συνειδητοποιήσει οι εταιρείε τη σημασία που έχει η ανείχνευση οποιασδήποτε προσπάθειας ε, κατάχρησης της ουσίας αυτής της προσπάθειας μας. Λοιπόν, έχουν ήδη οδηγήσει σε μείωση της κατάχρησης και η καλύτερη συνεργασία μεταξύ των αρχών μερικών κρατών μελών που μέχρι τούδε ενεργούσαν περισσότερο μεμονωμένα. Η γνωμοδότηση του, της υπηρεσίας προστασίας δεδομένων ε, μας έφτασε μόλις την προηγούμενη Παρασκευή. Μόλις λοιπόν προλάβαμε να την κοιτάξουμε στα γρήγορα, αλλά δεν νομίζουμε ότι μας δημιουργεί προβλήματα η γνωμοδότηση αυτή και η συγκήτρια είπε ότι θα προσέξει πολύ το θέμα αυτό. Θα συνεργαστούμε με την συγκήτρια και το Κοινοβούλιο λοιπόν ούτως ώστε να εντάξουμε τα διάφορα σημεία που αναφέρει η γνωμοδότηση. Διάφορα σημεία εξάλλου αφορούν ε, τα τεκτενόμενα στα κράτη-μέλη. Το Συμβούλιο λοιπόν επίσης που πήρε τη γνωμοδότηση θα πρέπει ε, να λάβει υπόψη αυτά τα σημεία. Πολλά σημεία επίσης αφορούν ε, τις διατάξεις για το εξωτερικό εμπόριο Είμαστε σε επαφή λοιπόν με την αρμόδια υπηρεσία της Κομισιόν και την καλέσαμε να αποτιμήσουμε από κοινού τα σημεία που αναφέρει αυτή η γνωμοδότηση της υπηρεσίας προστασίας δεδομένων. Και ένα σχόλιο που κάνει είναι αυτά τα κριτήρια ε, εξαίρεσης. Η τροπολογία που προτείναμε είναι αυτή που προτείνουμε και τώρα στον κανονισμό που ενεκρίθη μάλλον όχι εξαιρέσεων, είναι ε, οι διατάξεις που αφορούν την ε, απόρριψη κάποιας αίτησης ε, καταχώρησης στο Μητρό. Εάν όμως μπορούμε αυτήν την ισχύουσα που θέλουμε να επαναλάβουμε διάταξη και στον τροποποιημένο κείμενο να το διευκρινίσουμε, τότε να το εξετάσουμε. Σας διαβεβαιώ ότι ο τελικός κανονισμός θα είναι πλήρως ε, συμβατός με τις διατάξεις για την προστασία δεδομένων και ευχαριστώ. Θέλετε να κάνετε κυρία Κέλλερ και, άλλες, ε, και άλλα σχόλια. Μια που μιλάμε για στοιχεία. 33 τόνοι το 2009 ηρωίνης κατασχέθηκαν. Τι ποσοστό της, ε, του συνολικού εμπορίου οξικού ανιδρύτη είναι αυτό. Πολύ μικρό λέει η Κομισιόν. Το εμπόριο ανιδρύεται επίσης είναι πολύ μικρό. Η συνολική παραγωγή είναι περίπου ένα εκατομμύριο τόνοι όμικρον α ανιδρύτη. Στην Ένωση δεν έχω όλα τα στοιχεία απ' έξω, ε, παράγουμε περίπου το μισό. Τα στοιχεία υπάρχουν στην ε, μελέτη επιπτώσεων. Και το μεγαλύτερο ποσοστό της ουσίας όταν παράγεται καταναλώνεται εντός των εταιριών που το παράγουν. Και ένα μικρό ποσοστό ε, πωλείται σε άλλες εταιρείες και ένα ακόμη μικρότερο ποσοστό γίνεται αντικείμενο κατάχρησης. Αυτό που θα χρειαζόμασταν για να παραχθεί όλη η ηρωίνη που μας έρχεται από το Αφγανιστάν είναι περίπου 380-400 τόνοι ε, σε σχέση με το 1 εκατομμύριο που μόλις ανέφεραν. Αυτό καταδεικνύει ότι προσπαθούμε να ελέγξουμε ένα πολύ μικρό κλάσμα της συνολικής παραγωγής. Επαναλαμβάνω ότι το μεγαλύτερο τμήμα του παραγόμενου οξικού ανιδρύτη καταναλώνεται εντός των εταιριών που τον παράγουν. Ευχαριστώ. Και ο λόγος πάλι στην εισηγήτρια. Σας παρακαλώ και πάλι να βάλετε τα ακουστικά σας. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλευράς μου, όπως και τους σκιώδεις για τα σχόλια. Ιδίω τα ερωτήματα της κυρίας Καλέ ήταν πραγματικά πολύ εύστοχα και χρήσιμα για να ακούσουμε απαντήσεις. Τώρα εντάχει, μάλλον γρήγορα κι εγώ ε, θα προβώ σε ένα πρώτο σχέδιο έκθεσης, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε λίγες εβδομάδες. Αν λοιπόν οι σκιώδει ηγητέ θέλουν να μου δώσουν κάποιες ιδέες και προτάσεις, παρακαλώ να έρθουν σε επαφή μαζί μου το συντομότερο δυνατόν για να συμπεριλάβω τις απόψεις σας στο πρώτο σχέδιο. Και αν θέλουμε να περάσουμε τις τροπολογίες μέχρι τέλη ε, Φεβρουαρίου και να περάσουμε στην ψηφοφορία την έκθεση κάπου τον Απρίλιο στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, κάπως το χρονοδιάγραμμα κάπως έτσι δείχνει αυτή τη στιγμή, σας λέω λοιπόν και εγώ γρήγορα θα προβώ στην υποβολή του πρώτου σχεδίου έκθεσης. Παρακαλώ σκιώδες να έρθουν σε επαφή μαζί μου, ιδίω αν κάτι είναι πολύ σημαντικό για σας. Κατά τα λοιπά θα τα συζητήσουμε όταν θα έχετε λάβει το σχέδιο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ την κυρία Χέτ. Θα κλείσουμε εδώ τη συζήτηση για αυτό το σημείο για την τροποποίηση του κανονισμού για τις πρόδρομες ναρκωτικές ουσίες. Οπότε να προχωρήσουμε στο σημείο 11 της σημερινής διάταξης. Παρουσίαση τη Έκθεση 2012 σχετικά με τα ευρωπαϊκά δικαστικά συστήματα της ΣΕΠΕΣ, Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηλαδή, για την αποτελεσματικό δικαιοσύνη στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Θα έχουμε μια παρουσίαση που θα μας κάνει ο κ. Ζαν Πολζάν, πρόεδρος της ομάδας εργασίας ΣΕΠΕΣ ομάδα εργασία αξιολόγηση τη ΕΠΑΣ. Να τον καλωσορίσω. Σα ευχαριστούμε για την παρουσία σα. Σα ευχαριστούμε λοιπόν για τις παρουσίες στην Επιτροπή μας και την κυρία Τεκούρ και σα καλωσορίζω. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία μας να σας κάνετε σχετικά με δραστηριότητε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποτελεσματικότητα και ουσιανή Συμβουλή της Ευρώπης. Έχετε λοιπόν όπιον σα σε μια έκθεση η οποία εκπονείται κάθε δύο χρόνια, λαμβάνοντα υπόψη όλα τα δικαστικά συστήματα σχεδόν όλων των χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τελευταία έκθεση με ημερομηνία Σεπτέμβριο 2012 λαμβάνει υπόψη τα συστήματα 46 χωρών και καλύπτει ε, στον παρόδο και όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Θα δώσω λοιπόν τον το λόγο στον εισηγητή της έκθεσης, τον πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας Αξιολόγησης της ΣΥΠΙΤΣ, τον κύριο Ζαν Πολτζάν. Και μετά θα υπάρξει και κάποιος χρόνος για συζήτηση. Παρακαλώ και το λόγο. Jean Jean, je suis avocat général. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέγομαι Ζαν Πολτζάν, και είμαι πρόεδρος της ομάδας των εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης που ετοίμασαν αυτή την έκθεση. Τη γενική παρουσίαση θα την κάνει η κυρία Ντεκούρ που εκπροσωπεί το Συμβούλιο της Ευρώπης. Εγώ είμαι απλώς ένας ανεξάρτητος εμπειρογνώμων εκεί. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας εδώ στην Επιτροπή ΛΙΜΠΕ ΕΛΕΦ. Να σας πω πρώτα μερικά για το περιεχόμενο της έκθεσης γενικότερα και να σας, κάνω μερικές, να σας δώσω μερικές γενικές πληροφορίες για τη λειτουργία της ομάδας εργασίας αυτής του ΣΕΠΕΤΖ. Είναι για μας τιμή που σας παρουσιάζουμε εδώ τα αποτελέσματα των εργασιών μας αρχίσαμε πριν από έξι σχεδόν χρόνια και σας ξανά ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης της ΕΠΕΤΖΑ εορτάζει το 12, έορτασε το 12 τη δεκάτη επέτειό της γιατί ιδρύθηκε το 2002 για να προτείνει συγκεκριμένες και πρακτικές λύσεις χρησιμοποιήσιμες και από τα 46 χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης για να προωθηθεί η αποτελεσματικότερη εφαρμογή των νομικών εργαλείων που διαθέτει το Συμβούλιο της Ευρώπης για την καλύτερη οργάνωση της δικαιοσύνης, των προτύπων που καθορίζει δηλαδή, μετά για να φροντίσει τα πολιτικά προγράμματα που εφαρμόζουν τα δικαστήρια να λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες των χρηστών και τέλος για να συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων βρίσκοντας λύσεις πριν από την προσφυγή με επιφύλαξη βέβαια του άρθρου 6 της Σύμβασης. Για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες λοιπόν ισχύουν αυτά και εκεί έγινε μια αποτίμηση των αποτελεσμάτων των δικαστικών συστημάτων. Προτάσει, υποβλήθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης προς όφελος των πολιτών. Η ΣΕΠΕΣ λοιπόν κάθε δύο χρόνια κάνει μια αξιολόγηση των δικαστικών συστημάτων στην Ευρώπη, της καθημερινής λειτουργίας της δικαιοσύνης, δηλαδή στα κράτη αυτά. Πρόκειται για μια φωτογράφηση κάθε φορά της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης με πίνακες, γραφικές παραστάσεις που θα σας τις παρουσιάσει ο Ζαν Πολ σε λίγο και με συνοδευτικά σχόλια που μας βοηθούν να καταλάβουμε περισσότερο τα πράγματα. Τονίζουμε τις τάσεις που σημειώνονται στα δικαστικά συστήματα και ιδιαίτερα ταυτίζουμε τα προβλήματα για να τα λύσουμε για να βελτιωθεί η ποιότητα, η ισονομία της ε, υπηρεσίας, της δικαστικής υπηρεσίας. Επίσης συμβάλλουν στην αξιολόγηση αυτή, θέλουμε με την αξιολόγηση αυτή να βελτιώσουμε την αμοιβαία πληροφόρηση και γνώση για τη λειτουργία των συστημάτων ώστε να υπάρξει περισσότερη εμπιστοσύνη. Τέλος, καθορίζουμε έναν πυρήνα ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων που είναι ουσιώδης για να υπάρχει ίση μεταχείριση σε όλα τα κράτη-μέλη ώστε να υπάρξουν να καθοριστούν κοινοί δείκτες για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της δικαιοσύνης και για να φανεί αν πρέπει να εφαρμοστούν μεταρρυθμίσεις ή αν υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές. Στόχος της αξιολόγησης αυτής, της περιοδικής αυτής αξιολόγησης δεν είναι να γίνει μια ταξινόμηση των καλύτερων συστημάτων. Αυτό θα ήταν επιστημονικός απαράδεκτο. Απλώς επιτρέπει η αξιολόγηση της συγκρίσης μεταξύ χωρών μελών εφόσον είναι συγκρίσιμα τα συστήματα. Η διαδικασία λοιπόν βασιζόμαστε σε μια επιστημονική διαδικασία συλλογής, ανάλυσης, σύγκρισης δεδομένων. Η συλλογή βασίζεται σε πληροφορίες που υποβάλλουν τα κράτη-μέλη με βάση ένα ερωτηματολόγιο που αποστέλλεται κάθε δύο χρόνια στα Υπουργεία Δικαιοσύνης. Όλες οι εθνικές απαντήσεις λέγονται επαληθεύονται, καταγράφονται σε μια τράπεζα δεδομένων που έχει το, αυτή τη στιγμή πάνω από 3 εκατομμύρια στοιχεία. Επε, τα επεξεργαζόμαστε και τα αναλύουν οι εμπειρογνώμονές μας. Μετά συγγράφεται μια έκθεση που περιλαμβάνει και συγκριτικούς πίνακες και ανάλυση και εγκρίνεται στην Ολομέλεια της ΕΠΕΖ. Η έκθεση αφορά 46 χώρες μέλη, δηλαδή τις χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης εκτός από το Λιχτενστάιν. Και η τελευταία δημοσιεύτηκε το Σεπτέμβριο του 2012 και επισημοποιήθηκε από τη διάσκεψη των Υπουργών Δικαιοσύνη στη Βιέννη πέρυσι. Δούμε λίγα λόγια το γενικό πλαίσιο αξιολόγησης που κάνουμε και τώρα θα δώσω το λόγο στον Ζαν Πολ Ζαν που είναι πρόεδρος της ομάδας εργασίας που διαχειρίζεται την αξιολόγηση αυτή από την αρχή ήδη των εργασιών μας. Χάρη σε εκείνον υπάρχει η έκθεση και σημειώνονται βελτιώσεις και θα σας παρουσιάσει ορισμένες τάσεις που διαπιστώθηκαν από την τελευταία έκθεση στα ευρωπαϊκά δικαστικά συστήματα. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας παρουσιάσω ορισμένες γενικότερες τάσεις μετά από την παρουσίαση της κυρίας Δεβό. Σίγουρα θα έχετε διαβάσει τις 450 σελίδες της έκθεσης, σίγουρα, που αναλύουν 3 εκατομμύρια στοιχεία. Θα προσπαθήσω λοιπόν απλώς να σας παρουσιάσω μερικά κύρια θέματα που προκύπτουν από αυτήν. 46 χώρες σημαίνει πολλά εκατομμύρια κατοίκων, για, εκτός από το Λίχτενστάιν βέβαια, όλους τους κατοίκους των χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η έκθεσή μας έχει πάρα πολλά στοιχεία βέβαια και πολύ συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Η εφημερίδα Λεμόντα, ας πούμε, έγραψε δύο ολόκληρες σελίδες για να παρουσιάσει τα στοιχεία που ενδιαφέρουν τους Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης για την έκθεση αυτή. Αφορά τους προϋπολογισμούς της δικαιοσύνης, τις διορίες που προβλέπονται για την επεξεργασία θεμάτων διαζυγίων, τη θέση που έχουν οι χρήστες κλπ. Τον αριθμό των δικαστών που υπάρχουν ανακάτοικο, όλα τα βασικά στοιχεία για τα δικαστικά συστήματα συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση αυτή και κάθε φορά προσπαθούμε να τη βελτιώνουμε βέβαια με βάση δύο κύριους άξονες την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης και την ποιότητά της. Ενδιαφερόμαστε δηλαδή όχι μόνο για τις διορίες τους χρόνους διεκπαιρέωσης αλλά και το κόστος της δικαιοσύνης, τι χρησιμοποιείται ως ηλεκτρονικά μέσα και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Αυτό είναι που ενδιαφέρει κυρίως τα κράτη-μέλη. Μία πρώτη τάση που διαγράφεται από την έκθεση και που ενδιέφερε πολλούς είναι το ότι προσπαθούμε κάθε φορά, πέμπτη φορά γίνεται αυτό, τέταρτη που χρησιμοποιεί την ίδια μεθοδολογία, να βελτιώνουμε τους χρόνους διεκπαιρέωσης και τη βελτίωση της χρηματοδότησης, της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, στο νομικό σύστημα, τη θέση των χρηστών, τις εναλλακτικές λύσεις των διενέξεων και θέματα επιμόρφωσης των δικαστών, μισθών των δικαστών, αποζημίωσής τους για κάθε χώρα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο που χρησιμοποιούμε και θα προσπαθήσω να επανέλθω πιο λεπτομεριακά σε λίγο. Κάτι που ίσως επίσης σας ενδιαφέρει είναι ότι στο Συμβούλιο της Ευρώπης μου ζήτησαν το εξής. Έχουμε μια έκθεση λοιπόν για 46 ευρωπαϊκές χώρες τα 46 από τα 47 μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου ισχύει η Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και προσπαθούμε για πρώτη φορά να παρουσιάσουμε ορισμένα στοιχεία και γεϊκά για την Ένωση. Πρώτη φορά γίνεται αυτό. Και για ορισμένες υποψήφιες χώρες. <coughs> Γιατί συμπεριλάβουμε στοιχεία και για υποψήφιες χώρες της Ένωσης για να δούμε πώς λειτουργεί εκεί το δικαστικό σύστημα με την κυρία Ζουρή λοιπόν μια άλλη εμπειρογνώμονα του Συμβουλίου της Ευρώπης θα κάνουμε αυτά. για να διεκπαιρεώσουμε αυτά τα στοιχεία και την παρουσίασή τους. Λοιπόν, αρχίζω. Με μία μεγάλη γενική τάση στο σύνολο του Συμβουλίου της Ευρώπης για να δείτε τι ενδιαφέρει στις τελευταίες 4 χρήσεις 8 χρόνια, τα τελευταία 8 χρόνια δηλαδή σήμερα, όλες οι χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης έχουν ένα σύστημα νομικής βοήθειας, πράγμα που δεν ίσχυε πριν από 8 χρόνια. Με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση δηλαδή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οποιοδήποτε κατηγορείται ποινικό μπορεί σήμερα να έχει δωρεάν δικηγόρο σε όλες τις χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Άλλο ενδιαφέρον στοιχείο, η αύξηση του αριθμού των δικηγόρων και σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπου αυξάνεται ο αριθμός των δικηγόρων και η νομική αρρωγή. Και αυτό σημαίνει ότι το κράτος δικαίου έχει ακόμα μεγαλύτερη εφαρμογή από ό,τι πριν. Η Αντεκό μας είπε πριν ότι αρχίσαμε με 46 χώρες, το ίδιο σύστημα χρησιμοποιήσαμε και για τις 27 χώρες μέλη της Ένωσης. Δεν συγκρίνουμε όμως ασύγκριτα στοιχεία. Δεν συγκρίνουμε το Μονακό με τη Ρωσική Ομοσπονδία, ας πούμε. Δεν έχει νόημα, ούτε από άποψη πληθυσμού. Ούτε συγκρίνουμε ένα, μια πολύ φτωχή χώρα όπως την Αλβανία με μια πολύ πλούσια όπως η Γερμανία. Ούτε αυτό έχει νόημα. Προσπαθούμε λοιπόν να ομαδοποιήσουμε συγκρίσιμα στοιχεία με συγκρίσιμες καταστάσεις στις διάφορες χώρες, όπως χώρες της Ευρωζώνης με χώρες εκτός Ευρωζώνης. Επίσης, δεν θα συγκρίνουμε τα συστήματα για όλα τα θέματα, ας πούμε. Οι χώρες με εθνικό δίκαιο δεν μπορούν να συγκριθούν με χώρες σαν τη Γαλλία και την Γερμανία ως προς τον αριθμό των δικαστών. Δεν συγκρίνουμε λοιπόν το Ηνωμένο Βασίλειο με τη Γαλλία ή τη Γερμανία επ' αυτού γιατί 90% των υποθέσεων στις χώρες εθνικού δικαίου κρίνονται από μη επαγγελματίες δικαστές. Ιδού λοιπόν τα βασικά δεδομένα και οι πίνακες που έχουμε συγκρίνουμε χώρες με βάση τον πληθυσμό και τον λόγο του αέπανακάτοικο για να δούμε το σχετικό τους πλούτο και χρησιμοποιούμε τρία κριτήρια. Πληθυσμό, ΑΕΠ και μέσω ακαθάριστο ετήσιο μισθό. Τις υπόλοιπες λεπτομέρειες, της μεθοδολογίες δεν σας τις αναφέρω, αλλά ειδού τα αποτελέσματα του πίνακα για την Κροατία, επίσης μιλάμε στοιχεία για την Κροατία και για υποψήφιες χώρες όπως την Τουρκία, γιατί πιστεύουμε ότι είναι ενδιαφέρον να το δούμε και αυτό για το μέλλον. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε μία σύγκριση για το σύνολο των χωρών αυτών, για το ΑΕΠ, για τον πληθυσμό, για να δούμε ποιες χώρες είναι συγκρίσιμες. Και έχουμε εδώ και γραφικές παραστάσεις, ειδού οι χώρες της Ένωσης, βλέπουμε ότι η Γαλλία, η Γερμανία, δημογραφικά είναι πιο σημαντικές. Το ίδιο ισχύει και για τον εθνικό πλούτο. Από αυτά τα στοιχεία λοιπόν καταλήγουμε σε ορισμένα συμπεράσματα για τον πλούτο και τις επενδύσεις των χωρών στη δικαιοσύνη. Τι επενδύσεις γίνονται λοιπόν στη δικαιοσύνη. Ορίστε ένας άλλος πίνακας που έχουμε στα πλαίσια του Βουλής Ευρώπης εκπονήσει για τα 46 κράτη-μέλη. Αυτός ο πίνακας αφορά ευρώ ανακάτοικο, ανά 100.000 κατοίκους. Πόσα ευρώ από χώρα σε χώρα. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι η Γαλλία δίνει 60,5 ευρώ, ενώ η Πορτογαλία δίνει 64, η Ιταλία 65,9 κτλ. Έχουμε αυτό τον υπολογισμό σε ακαθάριστα ευρώ. Αλλά αυτό δεν λαμβάνει υπόψη ένα άλλο στοιχείο. Όταν μιλάμε για τον προπολογισμό της δικαιοσύνης, περί τίνος πρόκειται. Πρέπει να διευκρινίσουμε απόλυτα αυτό το σημείο για να μην υπάρξουν παρανοήσεις. Προϋπολογισμός της δικαιοσύνης, για να δούμε την αποτελεσματικότητα. Προϋπολογισμός της δικαιοσύνης μένει των δικαστηρίων, των δημοσίων αρχών, και της ε, δικαστικής αρρωγής. Αυτές είναι οι τρεις στήλε. Το άθροισμά τους το αποκαλούμε στη Γαλλία προϋπολογισμό των δικαστικών υπηρεσιών. Το πιο προφανές παράδειγμα όμως, ότι δεν είναι παντού έτσι. Στη Γαλλία ο προϋπολογισμός των φυλακών είναι εντός του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αλλά δεν το λαμβάνουμε υπόψη. Γιατί σε πολλέ χώρε ο προπολογισμό των φυλακών δεν είναι στον προπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνη. Συγκρίνουμε λοιπόν την ε, δικαστική συνδρομή, τα δικαστήρια και την εισαγγελία. Θέλουμε λοιπόν να δούμε τι σημαίνει προπολογισμό τη δικαιοσύνη για του πολίτε είναι ο προϋπολογισμός των ε, ε, δικαστικών υπηρεσιών και της δικαστικής συνδρομής ή αρρωγής, συγγνώμη, Και μετά θα εξετάσουμε επίσης ε, την πληροφορική, την επιμόρφωση των δικαστών κτλ. Προσθέτουμε και αυτά τα στοιχεία. Πρέπει να τα έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Εδώ λοιπόν τα έχετε, αλλά θα τα παρουσιάσω αναλυτικότερα αργότερα για τις χώρες μέλη και τις ε, υποψήφιες χώρες. Είναι λοιπόν αυτά τα σημαντικά στοιχεία. Εδώ βλέπουμε για παράδειγμα δύο τύπους ε, πίνακα. Βλέπουμε από τη μία τις ε, επενδύσεις που γίνονται για την, δηλαδή τις χρηματοδοτήσεις για τη ζώνη ευρώ και για την, τις χώρες που είναι εκτός ευρώ με βάση την ε, ισοτιμία του ευρώ την 1η πρώτου 2011. Οπότε πρέπει να λάβουμε υπόψη την διακύμανση άλλων ε, νομισμάτων όπως το πολωνικό σλότι. Πάνω με κόκκινο βλέπετε τους προπολογισμούς ε, των χωρών ευρώ, της ζώνης ευρώ. Βλέπετε η Ισπανία με κοκκινο βλεπετε τους προϋπολογισμούς των χωρων ευρω της ζωνης ευρω βλεπετε η ισπανια ειναι 99, συγγνώμη 91, η Γαλλία 60,5 κτλ. Ενώ αν κοιτάξουμε τις χώρες ε, που είναι με μπλε, οι αποκλήσεις είναι πολύ διαφορετικές, γιατί υπάρχουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις των ε, νομισματικών ισοτιμιών. Αυτά όμως είναι τα καθάριστα ποσά των προπολογισμών. Ποιος είναι όμως ε, ο πραγματικός προπολογισμό δικαιοσύνης. Εδώ τον έχετε. Δηλαδή, συγκρίνουμε τους προπολογισμού ε, για τη δικαιοσύνη σε σχέση με το ΑΕΠ. Η Πορτογαλία λοιπόν, εφόσον ε, έχει πολύ μικρότερο ΑΕΠ από την Γαλλία, στην ουσία δίνει πολύ περισσότερα. Αντίθετα, η Γερμανία δαπανά όσα περίπου και η Γαλλία, αλλά στην πραγματικότητα η Γερμανία επενδύει 100 όταν η Γαλλία δίνει μόνο 70 τόσα. Δηλαδή η Γερμανία επενδύει τελικά περισσότερα στη δικαιοσύνη. Και η Γαλλία επίσης ε, έχει μικρότερο ποσοστό, ποσό χρηματοδότησης της δικαιοσύνης από μια σειρά άλλες χώρες όπως η Ιταλία, η Ολλανδία κτλ. Δεν θα μπω τώρα στις λεπτομέρειες. Ένα μεγάλο τμήμα που είναι κίτρινο είναι η ε, μισθή. Βλέπετε το τμήμα της προφορικής επίσης, το κτηρίων για παράδειγμα. Ορίστε τα στοιχεία που βλέπετε. Η επιμόρφωση, η κατάρτιση των δικαστικών. Προσπαθούμε να ε, κάνουμε όλο και πιο συγκεκριμένα αυτά τα στοιχεία. Και εδώ έχουμε τους μισθούς, για παράδειγμα. Μισθοί των δικαστικών. Πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί ορισμένε χώρε του Συμβουλίου τη Ευρώπη με βάση αυτά τα στοιχεία, για παράδειγμα το Αζερβαϊτζάν, αύξησαν ε, του μισθού των δικαστικών, ενώ άλλε χώρε λόγω κρίση μείωσαν. Παράδειγμα η Πορτογαλία του μισθού των δικαστικών, όταν ε, μειώθηκαν οι μισθοί όλων των δημοσίων υπαλλήλων με βάση τα στοιχεία τα δικά μα προσάρμοσαν τους μισθούς των δικαστικών. Βλέπετε πόσο λεπτά είναι αυτά τα στοιχεία, πόσο μεγάλη επιρροή και συγκεκριμένοι έχουν. Τα στοιχεία τα έχουμε ως ακαθάριστους μισθούς, καθαρούς μισθούς, κάνουμε συγκρίσεις και έχουμε και αναλογίες σε σχέση με το μέσο μισθό κάθε χώρας ή το μέσο εισόδημα. Βλέπετε ότι για παράδειγμα ένας ε, δικαστής του δικαστηρίου κερδίζει 4,7 φορές το ε, μέσο εισόδημα του πληθυσμού, ενώ σε άλλες χώρες είναι πολύ περισσότερο αυτό. Ορίστε οι πίνακες που βλέπετε. Εδώ οι χώρες της Ένωσης, ορισμένες χώρες δίνουν πολύ μεγαλύτερους μισθούς σε σχέση με το μέσο εισόδημα των πολιτών Βεβαίως οι δικαστές ε, των ανωτάτων αγγλικών δικαστηρίων κερδίζουν πολύ περισσότερο γιατί είναι πρώην δικηγόροι που ε, γι' αυτό το λόγο προσλαμβάνονται. Κάτι άλλο που νομίζω ενδιαφέρει την Ένωση και όλα τα θεσμικά της όργανα, τι επενδύσεις γίνονται για τον εξυγχρονισμό του δικαστικού συστήματος. Για παράδειγμα για τις νέες τεχνολογίες της πληροφόρησης. Αν θεωρούμε ότι για να μειωθεί ε, ο χρόνος ε, μέχρι να αποδοθεί η δικαιοσύνη έχει μεγάλη σημασία ε, τι επενδύσεις γίνονται για να αξιοποιηθεί η μηχανοργάνωση. Συγκρίνουμε ένα χώρα και οι αναλύσεις μας εξετάζουν συγκριτικά τις επενδύσεις για την πληροφορική, για παράδειγμα υπολογιστέ, ένα δικαστικό, ένα ε, ε, βοηθητικό προσωπικό των ε, δικαστηρίων κτλ. Βεβαίως όταν θα υπάρξει αυτή η αναλυτικότερη έκθεση θα σας μεταβιβαστεί. Ορίστε ένας άλλος πίνακας που θεωρείται λεπτός για να συγκρίνουμε τις προσπάθειες που κάνει κάθε χώρα για να βοηθήσει τη δικαιοσύνη Πρέπει να δούμε ότι όσο πιο ψηλά είναι μια χώρα, τόσο πιο πλούσια είναι. Βλέπετε Λουξεμβούργο, Μονακό, Ελβετία. Και όσο πιο δεξιά είναι, τόσο περισσότερο επενδύει στη δικαιοσύνη της. Λοιπόν, πώς να σας το εξηγήσω τώρα. Θα προχωρήσω λίγο. οι χώρες στη μέση, Ολλανδία, Γερμανία κτλ. Αυστρία, Βέλγιο, Φιλανδία, χώρες με το ίδιο περίπου επίπεδο ΑΕΠ, όσο πιο δεξιά είναι, τόσο περισσότερο επενδύουν στη δικαιοσύνη τους. Χώρες με συγκρίσιμο λοιπόν ΑΕΠ, περισσότερο επενδύει η Σουηδία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Αυστρία, η Φιλανδία, η Γαλλία, ορίστε η ταξινόμηση μεταξύ συγκρισίμων χωρών. Δεν συγκρίνουμε όλες τις χώρες. Συγκρίνουμε μόνο συγκρίσιμες χώρες. Τώρα πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Να μια άλλη προτεραιότητα. Είχα πει ότι μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Τι τάσεις έχουμε εδώ. Απόλυτη προτεραιότητα. Δική μας και ξέρω και δική σας. Ορίστε ο πίνακας. Ευρώ αναπολίτη πόσο, ε, πόσα δίνουν στο σύστημά τους ε, δικαστικής αροχής. Βλέπουμε εδώ ότι οι αγγλοσαξονικές χώρες, Ηνωμένο Βασίλειο, συγκεκριμένα Σκοτία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Σουηδία, σε ευρώ δαπανούν περισσότερο. Θα πρέπει να το συγκρίνουμε και με την ευημερία της χώρας. Ορίστε λοιπόν για τις χώρες της Ένωσης προϋπολογισμός της δικαιοσύνης για την δικαστική αρρωγή. Εδώ βλέπετε ότι σε ευρώ οι χώρες που επενδύουν το περισσότερο είναι η Βόρεια Ιρλανδία, η Αγγλία, η Ολλανδία, 21, 21,6, η Σουηδία, η Ιρλανδία, η Φιλανδία, το Βέλγιο, η Γαλλία 5,4, Πορτογαλία 4,9 κτλ. Ορίστε οι χώρες. Η Αυστρία 2,2. Αυτό που ενδιαφέρει επίση. είναι όχι μόνο να δούμε πώς κατανέμουν τον προπολογισμό, σε κόκκινο είναι ο αριθμός υποθέσεων και το γκρι είναι το μέσο κόστος ανά υπόθεση. Αν μια χώρα δίνει πολλά για δικαστική συνδρομή, μήπως δίνει πολλά για λίγες υποθέσεις, πληρώνει πολλά τους δικηγόρους για παράδειγμα, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο όπου οι δικηγόροι μπάριστερ πληρώνονται με βάση το πραγματικό κόστος κάθε υπόθεσης ή δίνει για πολλές υποθέσεις όπως η Γαλλία ε, πληρώντας λίγο τους δικηγόρους σε περιπτώσεις για παράδειγμα η γαλλια πληρωνοντας πολλοί λαμβάνουν δικαστική αρρωγή για να έχουν πρόσβαση δικαιοσύνη και οι δικηγόροι παίρνουν λίγα και υπάρχει και τρίτη περίπτωση πολλές χώρες με δικηγόρους που αμείβονται καλά. Ολλανδία. Τεράστιο κόστος δικαστικής αρρωγής και ξέρω ότι συζητείται ρύθμισή του. Πολλοί έχουν έτσι πρόσβαση μέσω της δικαστικής αρρωγής δικαιοσύνη και οι δικηγόροι επίσης έχουν από το υψηλότερο κόστος ε, αμοιβή ανά υπόθεση στην Ευρώπη. Άλλο οικονομικό που θεωρώ σημαντικό είναι η πρόσοδη της δικαιοσύνης. Δηλαδή πρέπει να πληρώσουμε και φόρους εκτός από το δικηγόρο μας. Με το 2010 μόνο δύο από τις 46 χώρες είχαν δωρεάν δικαιοσύνη, Λουξεμβούργο και Γαλλία. Από το 2011 υπάρχει ένας φόρος και για τη δικαιοσύνη, μόνο στο Λουξεμβούργο είναι δωρεάν η πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Πιο σημαντικό το κόστος είναι στην Αυστρία, τη Μαλτία, τη Σερβία, τη Γερμανία σε σχέση με τα έσοδα της δικαιοσύνης. Γιατί τα έσοδα της δικαιοσύνης τα υπολογίζουμε στους προπολογισμού. Τώρα απλώς θα σας δείξω μερικούς πίνακες, μερικά παραδείγματα δηλαδή, του τι κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Παράδειγμα, ο αριθμός δικαστών αναχώρα, επαγγελματιών δικαστών. Γι' αυτό κάνω την ε, διευκρίνηση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο 3,6 δικαστές επαγγελματίες. Αλλά, όπως σας είπα, δεν ε, λαμβάνουμε υπόψη του magistrates που δεν είναι επαγγελματίε. Γερμανία 24,3 είναι το, πιο, ε, το σύστημα που έχει του περισσότερου επαγγελματίε δικαστέ. Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία είναι γύρω στο 10 ανά 100.000. Στη Γαλλία οι εμπορικοί ε, δικαστές για εμπορικά θέματα και οι ειρηνοδίκες πολλές φορές δεν είναι επαγγελματίες. Δηλαδή οι δικαστές για ε, μικρή σημασία υποθέσεις. Επίσης λαμβάνουμε υπόψη και τους δικαστικούς υπαλλήλους. αναπολίτες. βλέπουμε ότι είναι μεταξύ 2, 3, 5. Όσο περισσότεροι δικαστικοί υπάλληλοι υπάρχουν στο σύστημα, τόσο πιο σκούρο είναι το χρώμα στον πίνακα αυτό. Βλέπουμε λοιπόν στην Ανατολική Ευρώπη έχει μικρότερους ε, αριθμούς. Αν κάνουμε ένα πίνακα για τις 27 χώρες, στο πράσινο έχει τον αριθμό δικαστών και στον κρήτο τον αριθμό δικαστικών υπαλλήλων. Βλέπετε τα συστήματα που για 100.000 κατοίκου έχουν περισσότερους ή λιγότερους ε, δικαστές. Στο πάνω μέρος είναι Μοντενέγρο, Σλοβενία, Κροατία, Μακεδονία, λέει ο μιλητής, χώρες της πρώην Ιουκοσλαβίας. Έχουν τους περισσότερους δικαστές και οι υπαλλήλου των δικαστηρίων. Και η Πολωνία, η Τσεχία κτλ. Έχουμε επίσης και το ποσοστό βοηθών του δικαστή, ένα δικαστή. Ε, αν έχετε ερωτήσεις, θα επανέρχομαι. Επίσης, ε, μελετήσαμε και τον αριθμό εισαγγελέων. Διαχωρίζουμε τους εισαγγελεί από τους δικαστές. Νομίζουμε πως είναι πολύ σημαντικό. Αλλά ο αριθμός λοιπόν εισαγγελέων διαπιστώνουμε ότι είναι περισσότεροι στη Γερμανία από ότι στη Γαλλία, περισσότεροι στην ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο η υπηρεσία ε, εισαγγελέων του ε, στέματος Crown Prosecution Service. Απλώς όμως ε, είναι η διαφορά μεταξύ των δύο συστημάτων ε, έχει πολύ διαφορετικό ρόλο λοιπόν η εισαγγελία σε συστήματα από άλλα. Η εισαγγελία σε ορισμένα συστήματα περνάει πολύ πιο εύκολα σε απαγγελία κατηγοριών από ότι σε άλλα που γίνονται πολύ περισσότερε ανακρίσεις. Επίσης, σε ορισμένες χώρες οι δυνατότητες ε, έφεσης και άλλων προσφυγών είναι πολύ πιο περιορισμένες από άλλες. Για παράδειγμα, στη Γαλλία οι εισαγγελείς έχουν πάρα πολύ δουλειά και είναι ιδιαίτερα ολιγάριθμοι, γιατί έχουν πολύ εκτεταμένες αρμοδιότητες. Κάτι άλλο που ενδιαφέρει είναι Επίσης, ε, ο λεγόμενος, ε, η λεγόμενη γυάλινη ή αόρατη οροφή. Τι ποσοστό είναι γυναίκες. Για πρώτη φορά αναφέρουν τέτοια στοιχεία. Βλέπετε λοιπόν την κατανομή αναφύλο. Γκρι είναι ο αριθμός των δικαστών. Μάλλον μόβι είναι οι γυναίκες σε μοβ και πράσινο οι άνδρες. Θα δείτε λοιπόν ότι τις περισσότερες γυναίκες τις έχουν η Σερβία, Ρουμανία Λετωνία, Σλοβενία. Και λιγότερες γυναίκες δικαστές είναι στη Σκοτία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία κτλ. Τα συστήματα common law, όπου οι άνδρες είναι 75 με 80%. Βλέπουμε λοιπόν τι προσπάθειες πρέπει να γίνουν ακόμη ε, για να προσληφθούν ε, περισσότερες γυναίκες. Ισορροπία βλέπουμε στη Γαλλία, την Αυστρία, την Ιταλία, όπου είμαστε περίπου στο 50-50. Γενικά στο σύστημα δικαιοσύνης. Και οι προσλήψεις ε, είναι όλο και περισσότερο γυναικών. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, 75% των ε, νέων δικαστών είναι γυναίκες. 75%. Αυτό επίσης καταδεικνύει ότι οι γυναίκες είναι ε, στο κάτω μέρος της ε, πυραμίδας και οι άντρες είναι στην κορυφή. Να για όλα τα δικαστήρια. Λευκό είναι οι γυναίκες πρόεδροι δικαστηρίων. Μόνο στην Ελλάδα λοιπόν, την Πολωνία, την Κροατία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία οι γυναίκες ε, πρόεδροι δικαστηρίων πρωτοβαθμίων είναι περισσότερες από ότι οι άνδρες. Μόνο πέντε από τις 27 χώρες της Ένωσης. Ενδιαφέρον στοιχείο νομίζω αυτό. Και εδώ βλέπετε τα στοιχεία επίση για τα εφετεία, τα ακυρωτικά δικαστήρια κτλ. Τώρα για τους εισαγγελεί. Είναι χειρότερα ακόμη τα πράγματα στην περίπτωση των εισαγγελέων. Ακόμη περισσότεροι άνδρες από ό,τι γυναίκες. Και λιγότερες γυναίκες ε, σε επικεφαλής εισαγγελιών. Δικηγόροι τώρα στις διάφορες χώρες η τάση που προανέφερα, βλέπετε εδώ αυτή την καμπύλη, και αυτό είναι ενδιαφέρον, μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις για τρεις περιόδους αναφοράς. Τα στοιχεία λοιπόν που συλλέξαμε το 2006, 2008 και 2010. Η τάση λοιπόν που βλέπουμε είναι να αυξάνονται οι δικηγόροι και ιδίω στην Ανατολική Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι αναπτύσσεται το κράτος δικαίου σε αυτές τις χώρες. Με βάση λοιπόν τις τρεις περιόδους αναφοράς φαίνεται ποιες είναι οι χώρες με τους περισσότερους δικηγόρους ανακατοίκους. Ιδού οι χώρες αυτές είναι με πιο σκούρα χρώματα φυσικά οι χώρες του Νότου. Οι τέσσερις χώρες που έχουν τους μεγαλύτερους αριθμούς δικηγόρων ανακατοίκους Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία, Μάλτα. Διότι η λειτουργία του συστήματος δικαιοσύνης δίνει πολλές εξουσίες, ιδίως στο αστικό δίκαιο, στους δικηγόρους. Κάνουμε επίσης και κάποιες μελέτες για τους, τις υποθέσεις που καθυστερούν και το χρόνο εκδίκασης. Αυτά τα στοιχεία νομίζουμε πως είναι πολύ ενδιαφέροντα. Αυτές τις αναλογίες τις βλέπετε και για την Ένωση συνολικά, μεταξύ αριθμού δηλαδή δικηγόρων, με βάση τον ορισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης, αυτοί που μπορούν να εκπροσωπήσουν τους ε, διαδίκους και οι δικηγόροι ανά επαγγελματίες δικαστές. Περισσότεροι δικηγόροι ανά δικαστές βεβαίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό είναι φυσιολογικό. Και αμέσως μετά είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Αλβανία. Πολύ σημαντική αυτή η αναλογία γιατί δείχνει τον φόρτο εργασίας των δικαστών. Θα περάσω πολύ γρήγορα τώρα μερικές ε, σελίδες για να περάσω στις ερωτήσεις απαντήσεις. Πέντε λεπτά ακόμη. Αποτελεσματικότητα και ποιότητα της δικαιοσύνης σε σχέση με όλη αυτήν την χρηματοδότηση και προσπάθεια. Πρώτο στοιχείο. Γίνονται πολλές μεταρρυθμίσεις σε πολλές χώρες. Υπάρχουν πολλά ή λίγα δικαστήρια ανακατοίκους. Δικαστήρια γεωγραφικά κατανεμημένα. Πολύ σημαντικές διαφορές από χώρα σε χώρα. Εξαρτάται από διάφορα θέματα βέβαια. Δεν θα συγκρίνουμε για παράδειγμα την Γαλλία με Ολλανδία. Έχει να κάνει με την έκταση τη χώρα και τον αριθμό των κατοίκων. Αλλά υπάρχει μια τάση μείωση των δικαστηρίων ούτω ώστε να είναι πιο αποτελεσματικά στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων που γίνονται. Στις, ε, όλα αυτά στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης ενώ στην Ανατολική Ευρώπη έχουμε το αντίθετο. Λόγω ανάπτυξης του κράτους δικαίου επανερχόμεθα σε δικαστήρια που είναι κοντά στον πολίτη. Συγκρίνουμε επίση την ανάπτυξη τη πληροφορική σε διάφορε χώρε, μια σειρά από δείκτες. Όσο πιο σκούρα είναι η χώρα, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η πληροφορική, τόσο περισσότερε επενδύσει έχουν γίνει στον τομέα αυτό. Για παράδειγμα, ανάπτυξη βίντεο διασκέψεων, τηλεδιασκέψεων, στην ε, ποινική δικαιοσύνη για να γίνονται εξοικονομίες χρημάτων. Οι μπλε χώρε έχουν τέτοιο σύστημα τηλεδιασκέψεων, προσπαθούν να λύσουν τα δεδομένα. Ενδιαφέρει πολύ ε, το θέμα αυτό. Ε, επίσης ενδιαφέρει ε, το σύστημα διαμεσολάβησης ή διαιτησίας για αστικά ή ποινικά θέματα. Εδώ έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές στα συστήματα διαιτησίας, γιατί οι ορισμοί είναι πολύ διαφορετικοί είναι δικαστική διαμεσολάβηση, έξω δικαστική που διατάσσεται από το δικαστή, δωρεάν, ε, που κοστίζει κτλ. Δύο σαφείς δείκτες είναι διεθνείς, τους οποίους ακολουθούμε και σε εθνικό επίπεδο και για κάθε δικαστήριο. Πρώτα απ' όλα ο ρυθμός εκδίκασης και επίσης ο χρόνος που χρειάζεται για να εκδικαστεί κάθε υπόθεση. Λοιπόν, ε, αυτός ε, ο, ο πρώτος δείκτης που είναι ο δείκτης ε, ε, εκδίκασης έχει να κάνει με το εάν για κάθε εκδίκαση 100 υποθέσεων προστίθεται πάνω από 100 ή όχι. Και ο δεύτερος δείκτης, ο χρόνος για την εκδίκαση, τι χρόνος χρειάζεται για να αντιμετωπιστούν οι εκκρεμούσε παλιέ υποθέσει. Συγκεκριμένα παραδείγματα αστικού δικαίου, εμπορικού δικαίου, κατά τη δικία και όχι, για να δούμε ποιο είναι ο μέσος χρόνος για τις κατά τη δικία. Για παράδειγμα, στην Ανατολική Ευρώπη θα δείτε ότι εκτός από τη Ρωσία που τα κάνει διαφορετικά, έχουμε περισσότερο χρόνο και θα επανέλθω για τις χώρες της Ένωσης για κάθε χώρα. Λοιπόν, έχουμε τα στοιχεία για τις κατά αντιδικία, χωρίς αντιδικία. Η Ιταλία έχει πολύ καλό αποτέλεσμα, αντίθετα από ό,τι θα περίμενε κανείς, διότι το 2010 είχαν πολλές εκκρεμούσες υποθέσεις, γιατί δεν λειτουργεί σωστά η δικαιοσύνη, αλλά το 2010 άρχισε να εφαρμόζεται ένα σύστημα απλούστευση των υποθέσεων που επέτρεψε να εκδικαστούν πολλές Λειτουργεί αρκετά καλά αυτή η μεταρρύθμιση. Μετά έχουμε διάφορε υποθέσει για παράδειγμα, για τι τρει περιοδου αναφορά διαζύγια κατά τη δικία. Μετρήσαμε το χρόνο εκδίκαση αυτών των διαζυγίων σε διάφορε χώρε. Αριθμός ημερών, για παράδειγμα, περισσότερε στην Ιταλία. 538 ημέρε. Πρωτοδίκω για μια κατά δική υπόθεση διαζυγίου. Ορίστε λοιπόν παραδείγματα για να μπορέσει να τροφοδοτηθεί η συζήτηση. Υπάρχουν πολλά στοιχεία. Ε, βέβαια, σε 450 σελίδες ο καθένας πρέπει να δει τι τον ενδιαφέρει και να δει πώς συγκρίνονται τα συγκρίσιμα. Η εργασία μας αυτή θα παρουσιαστεί σε μερικούς μήνες. Μπορεί οπωσδήποτε να σας βοηθήσει να εξάγεται δηλαδή από τα δεδομένα μας ε, τα στοιχεία που αφορούν τις 27 χώρες μέλη και τις υποψήφιες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ζώ για την εξαιρετική, πραγματικά εξαιρετική αυτή παρουσίασή σας. Ήταν λίγο μακροσκελής βέβαια, αλλά άξιζε τον κόπο. Ήταν λεπτομερής, ενδιαφέρουσα και πολύ σημαντική θα έλεγα. Τον υπόλοιπο χρόνο μας θα ακούσουμε παρατηρήσεις, σχόλια και απορίες των μελών της Επιτροπής μας. Και εγώ ε, είμαι υπεύθυνος για την έκθεση της Στοκχόλμης. Μήπως όμως θα μπορούσατε να μας δώσετε και τους δίσκους, τα CD με τα στοιχεία. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Αν δεν έχεις εντέσει, στικάκι. Και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να δώσουμε συνέχεια σε αυτά τα συμπεράσματά σας. Πρέπει να διαδοθούν όλα αυτά, να μαθευτεί δηλαδή και να ασχοληθεί και η ίδια η Κομισιόν. Scoreboard το λένε αυτό για τη δικαιοσύνη. Αξιολόγηση δηλαδή για την αποτελεσματικότητα και ποιότητα των δικαστικών συστημάτων. Ιδιαίτερα για τα 28 28 επαναλαμβάνω μέλη της Ένωσης για να συμπληρωθεί έτσι η δουλειά σας με τα δικά μας στοιχεία. Τώρα, θα δώσουμε το λόγο σε δύο μέλη που τον ζήτησαν. Μπερί Τσίπελ πρώτη. Ευχαριστώ. Δεν είχα ακόμη δυνατότητα, δυστυχώς, να βάλει τα ακουστικά του ο κύριος Ζω. Εντάξει. Δεν πρόλαβα λοιπόν ακόμη να διαβάσω λεπτομερώς την έκθεση. Ευχαριστώ λοιπόν για την αναλυτική παρουσίαση. Όπως και στο παρελθόν, τα στοιχεία αυτά θα μας βοηθήσουν πολύ για τις συζητήσεις μας. Θα είναι μια πολύ πολύτιμη βάση οι διαφορές των ε, συστημάτων απονομής δικαιοσύνης. Για τέσσερα σημεία να υποβάλω ερωτήσεις. Μιλήσατε για την δικαστική αρρωγή που υπάρχει τώρα πλέον σε όλες τις ε, χώρες μέλη. Αναφέρατε στοιχεία. Θα με ενδιέφερε εάν υπάρχουν μεγαλύτερες διαφορές όσον αφορά τις προϋποθέσεις χορήγησης της ε, δικαστικής ε, συνδρομής αυτής, αρρωγής, συγγνώμη. Υπάρχουν ε, συγκεκριμένοι κανόνες για το πότε έχει δικαίωμα κανείς. Δεύτερον, κατάρτιση των δικαστών. Αναφερθήκατε στο κόστος ανακράτος. Υπάρχουν διαφορές για το είδος της κατάρτισης των επαγγελματιών. Έχουμε μια συνολική εικόνα για το εάν έχουν τέτοια δυνατότητα κατάρτισης όλοι οι δικαστές και σε τακτά χρονικά διαστήματα ή είναι δύσκολο να έχουμε τέτοια στοιχεία. Τώρα, για τους προπολογισμού της δικαιοσύνης, για πληροφορική. Υπάρχουν, είπατε, διαφορετικά συστήματα για την ποινική και αστική δικαιοσύνη. Έχετε πληροφορίες για, το εάν, για τον εξυγχρονισμό, την μηχανοργάνωση, δαπανώνται περισσότερα στον α ή στο β τομέα. Και είπατε αναλυτικά ε, ποια είναι τα στοιχεία που έχετε για τους δικαστές, τους δικηγόρους, τους δικαστικούς υπαλλήλου. Συνολικά για τους απασχολούμενους στα συστήματα δικαιοσύνης, θεωρείτε ότι ο αριθμός των απασχολουμένων έχει σχέση με την ποιότητα της δικαιοσύνης. Οι χώρε που έχουν μεγάλο ρυθμό απασχολημένων στη δικαιοσύνη ε, διευκολύνουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, έχουν αποτελεσματική δικαιοσύνη. Να αρκεστώ σε αυτά, ελπίζω ε, να λάβω ενδιαφέρουσε απαντήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τι ερωτήσει σα. Ο κύριος Μπρόγκ. Ευχαριστώ. Και ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρησή μου σε άλλη επιτροπή, οπότε μπορεί κάτι να έχασα. Έχετε κάνει κάποια σύγκριση ανάμεσα στον αριθμό των ποινικών διώξεων ανά 100.000 ας πούμε ε, πληθυσμού. Γιατί σε κάποιες χώρες είναι πιο πιθανό να βλέπουμε τέτοιες ποινικέ διώξεις από τις άλλες χώρες. Αυτό βεβαίω μπορεί να οφείλεται σε διαφορετικό επίπεδο κλιματικότητα, από χώρα σε χώρα ή ε, κάποιες χώρες αρέσκονται να κάνουν τις ποινικές διώξεις. Έπειτα, έχετε παρατηρήσει σημαντικές διαφορές ανάμεσα στον αριθμό αγωγών ε, που ανά 100.000 κατοίκους. Δηλαδή χώρες που δείχνουν να προσφεύγουν σε δικαιοσύνη πιο πολύ από άλλους. Αναφερθήκατε και στη διαμεσολάβηση ή διαιτησία. Γενικότερα στις εναλλακτικέ μεθόδους ε, επίλυση διαφορών. σε κάποιες περιπτώσεις ε, μιλάμε για τη διατησία αυτής εξ αρχής ή είναι συνέπεια άσκησης μιας αγωγής. Και κατά πόσον αυτέ οι εναλλακτικέ μέθοδοι επίλυση διαφορών είναι πραγματικά αποτελεσματικέ, ώστε να μην δαπανώνται και πάρα πολλά χρήματα ε, στα δικαστήρια. Euh, απαντήσω πολύ σύντομα προς τον πρόεδρο. Ναι, στην ιστοσελίδα της ΕΠΕΣ στο Συμβούλιο της Ευρώπης έχετε όλα τα στοιχεία. Είναι προσβάσιμα και της έκθεσης και αναχώρα όλες οι απαντήσεις που έδωσαν οι χώρες σε μορφή PDF. Έχουμε και άλλους συνεργάτες και ερευνητές για συγκεκριμένα θέματα, αλλά εμείς ελέγχουμε το σύνολο της μεθοδολογίας των δεδομένων, γιατί εδώ μιλάμε για δεκαετή δουλειά των συνεργατών μας. Δεν θέλουμε λοιπόν να γίνουν πρόχειρες και βιαστικές ερμηνείες των δεδομένων αυτών, αλλά επεξεργασία τους με επιστημονικό τρόπο και με όλες τις μεθοδολογικές εγγυήσεις που χρειάζονται. Και οι εγγυητέ είναι ακριβώς η ομάδα των εμπειρογνωμόνων από όλες τις χώρες. Για την κυρία τώρα, για το πρώτο, Πράγματι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο θέμα της αρρωγής. Έχουμε εδώ συγκεκριμένα στοιχεία αναχώρα. Αν έχει αποφευθεί ή όχι η δίκη, αν ο δικαστής αρχολήθηκε κτλ. Δεν μπορώ να σας πω όμως γενικά. Δεύτερον, για την εκπαίδευση. Χωρίζουμε, διαχωρίζουμε την αρχική εκπαίδευση από την ειδίκευση και αυτό αναχώρα και με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Πάρα πολύ συγκεκριμένα. Και τέλος, για κάθε θέμα έχουμε και τα εκρεμή θέματα ή ερωτήσεις ανοιχτές όπου κάθε χώρα παρουσιάζει τα προβλήματα που βλέπει. Για την επένδυση σε νέες τεχνολογίες έχουμε τρία επίπεδα ανάλυσης η άμεσ, το άμεσο υλικό που χρησιμοποιεί ο δικαστής και η βοηθή του ή το γενικότερο σύστημα. Και εδώ υπάρχουν λεπτομερή στοιχεία. Και τέταρτο ερώτημα, πολύ σημαντικό, όχι. Δεν λειτουργούν καλύτερα τα δικαστικά συστήματα με το περισσότερο προσωπικό. Καμιά φορά το αντίθετο, γιατί μπορεί το πολύ προσωπικό να δημιουργεί πολύ γραφειοκρατία. Πρέπει να εξετάσουμε συγκεκριμένα τα αποτελέσματα. Οι χώρες που επενδύουν περισσότερο δεν έχουν αναγκαστικά τα καλύτερα αποτελέσματα. Μπορώ να δώσω και παραδείγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ας μην το κάνω για να μην ε, κατηγορήσω μια χώρα που όλοι υπονοείται. Ο κύριος Μπρόντς, τα ποινικά στοιχεία είναι πολύπλοκα, γιατί είναι διαφορετικά τα δικαστικά συστήματα και δεν υπάρχουν οι ίδιες ποινικέ κατηγορίες. Υπάρχει ένα source book ευρωπαϊκό για τις ποινικέ αυτές κατηγορίες. Άλλο crime, άλλο misdemeanor ας πούμε. Πλημέλημα, έγκλημα, παράπτωμα κτλ. Αλλά τα έχουμε και αυτά όλα τα στοιχεία ανάλογα με τον αριθμό των κατοίκων ανά 100.000. Αλλά Στη Γερμανία ας πούμε υπάρχει πολύ διοικητική επεξεργασία των ποινικών υποθέσεων, στην Ολλανδία με άλλο τρόπο το διεκπεραιώνουν. Και τέλος, ναι, είμαστε υπέρ του συστήματος της διαμεσολάβησης και της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Θέλουμε να επεκταθούν τέτοια συστήματα και προσπαθούμε να το πουλήσουμε σε εισαγωγικά αυτό και στις χώρες μέλη. Αλλά και εδώ υπάρχουν πολύ διαφορετικά συστήματα όταν εφαρμόζονται τέτοιες εναλλακτικέ επιλύσεις. Όσο για τις σχέσεις μας με την Κομισιόν, προσπαθήσαμε να καταρτήσουμε ένα scoreboard για την Κομισιόν, τη αιτήση της. Για το πρώτο σας ερώτημα, συνεργαστήκαμε πέρυσι με την Κομισιόν για τη χρησιμοποίηση των δεδομένων αυτής της αξιολόγησης σε μια μελέτη για την επίπτωση της λειτουργίας των δικαστικών συστημάτων στην δημοσιονομική κατάσταση των χωρών. Αρχίζει λοιπόν μια τέτοια συνεργασία και φυσικά θα συνεχιστεί ακόμη όμως προσπαθούμε να δούμε πώς θα μπορούσε να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Κομισιόν ΔΕ είναι παρατηρήτρια σε όλες μας τις εργασίες και συνεδριάσεις. Κυρία Δεκό, κύριε Ζαν, σας ευχαριστούμε και σας συγχαίρουμε για την ποιότητα των ερευνών σας, του ομάδας εργασίας σας και για την ποιότητα της παρουσίασής σας βέβαια. Νομίζω θα παραμείνει στα χρονικά και θα είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο για την Επιτροπή ΕΛΕΦ, ΛΙΜΠΕ, για την ανάλυση και για τις πρωτοβουλίες που μπορεί να χρειαστεί να αναλάβουμε για τη βελτίωση των δικαστικών συσουτημάτων και για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών στην Ένωση. Σας ευχαριστώ εκ νέου. Θα συνεχίσουμε στις 3. Στις 3.